εκλογή του κυρίου Έντουαρτ Τσέζακ που αντικαθιστά τον κύριο Αντρέι Ντούντα από τις 11 Ιουνίου 2015. Το Κοινοβούλιο καταγράφει την εκλογή του κυρίου Τσέζακ, τον καλωσορίζω και θυμίζω ότι ε, συμμετέχει στο Κοινοβούλιο με όλα τα δικαιώματα και στα όργανα βέβαια του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από το κανονισμό Στη συνέχεια της παρέτησης του κυρίου Εμμανουήλ Γλέζου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει την ε, κενότητα της θέσης του από τις 8 Ιουλίου 2015 σύμφωνα με το κανονισμό και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Μετά από την παρέτηση της κυρίας Μάριτ Πάουλσεν, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την ε, θέση του και που ισχύει από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 σύμφωνα με το κανονισμό και ενημερώνει τις ε, αρμόδιες εθνικές αρχές. Σας ενημερώνω επιπλέον ότι η Νομική Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 16 Ιουνίου 2015 προέβη στην